Liebe Kolleginnen, Kollegen, guten Morgen. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτική μας Επιτροπής. Είχαμε τη συνάντηση των συντονιστών πιο πριν. Και γραπτά θα υποβληθούν οι αποφάσεις μας εκεί στη συνάντηση των συντονιστών. Θα τις πάρετε γραπτά. Τώρα έχουμε το σημείο 16 στην ημερησία διάταξη. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρατήρησης της ε, Γης, ε, GMES. Και έχουμε τον Βιτόριο Πρόντι που έχει αναλάβει τη σύνταξη αυτής της έκθεσης ως εισηγητής. Μια γνωμοδότηση είναι από πλευρά μας για την Επιτροπή Ήτρε. Ο Βιτόριο Πρόντι θα κάνει την εισαγωγή λοιπόν, θα παρουσιάσει την έκθεση του. Παρακαλώ Πρόντι. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς που μου εμπιστευθήκατε την σύνταξη αυτής της ε, έκθεσης και έχω να σας πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά αυτήν την ε, παρατήρηση, την εποπτεία για το περιβάλλον και για την ασφάλεια. υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί λόγοι για τους οποίους γίνεται πάρα πολύ ε, κρίσιμη αυτό το νομοθότημα και πρέπει να σας ε, ε, τονίσω ότι αυτό το σχέδιο πρόκειται να ενταχθεί στο πλαίσιο της ε, σημερινής πολιτικής παρατήρησης του διαστήματος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και επομένως έχουμε μια σειρά ε, τοπικών πρωτοβουλειών που σχετίζονται με αυτήν την ε, γενικότερη, την σφαιρικότερη. Όλα είναι και περισσότερο θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε διάφορες πληροφορίες, διάφορα δεδομένα που έχουν σχέση με το, διάλειμμα, γιατί, με το διάστημα, συγγνώμη, διότι ε, μεταβάλλονται όλα τα δεδομένα κυρίως όσον αφορά το κλίμα. Όμως πέραν αυτού χρειαζόμαστε το να συλλέξουμε δεδομένα τα οποία ε, όλο ένα και μεγαλύτερη ποικιλία εμφανίζουν. Επομένως, το πρόγραμμα GMES είναι μια πρωτοβουλία πάρα πολύ χρήσιμη για την παρατήρηση του διαστήματος αλλά και του περιβάλλοντος και της ασφάλειας γενικότερα. το GMS, κινείται γύρω από το εισάξονες, πρωτα πρώτα-πρώτα παρακολούθηση του διαστήματος. Δεύτερον, υπάρχει η δυνατότητα μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος να βοηθήσουμε ούτως ώστε να έχουμε ε, καλύτερες τεχνολογίες παρατήρησης και παρακολούθησης. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Και σας ε, υπενθυμίζω ότι μεταξύ άλλων θα μπορέσουμε να παρατηρούμε με, ε, και να μελετούμε διάφορες παραμέτρους που μέχρι σήμερα δεν είχαν ληφθεί υπόψη, δεν είχαν επισημανθεί όπως η θερμοκρασία της επιφανείας ή το επίπεδο των ωκεανών. Αυτό γιατί τώρα θα μπορέσουμε να παρακολουθούμε πολύ καλύτερα από ό,τι πριν, κάτι το οποίο επιβάλλεται να γίνεται. Επίσης, ε, το αλάτι στη θάλασσα. Και αυτό τώρα θα μπορούμε να το μετρούμε καλύτερα, που είναι πολύ σημαντικό γιατί με τη σειρά του ε, έχει να κάνει με το επίπεδο της θερμοκρασίας του πλανήτη. Επίσης, μπορούμε τώρα να προβούμε σε μέτρηση της ε, υγρασίας, κάτι το οποίο επίσης σχετίζεται με την μέτρηση της ε, συνολικής χλωρίδας του πλανήτη. Επίσης θα μπορούμε να παρακολουθούμε και την κατάσταση των ερήμων. Με αυτό το πρόγραμμα θα έχουμε έναν συντονισμό ε, μέτρων που ήδη ε, έχουν ληφθεί και αφορούν οι ωκεανούς και επιφάνεια της γης. Και όπως είδαμε στη σχετική οδηγία που φορούσε τις πλημμύρες. Σας επενθυμίζω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε αυτές τις πληροφορίες από το διάστημα με μετρολογικά δεδομένα για προβλέψεις μέσο και μάκρο πρόθεσμες. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε έτσι βήματα πρόοδο όσον αφορά την πρόβλεψη κάποιων θεομηνιών. Επίσης, μπορούμε να συνδυάσουμε την χρήση δορυφόρων με την χρήση των ραντάρ και άλλων επιγείων σταθμών παρακολούθηση. Όλα αυτά μας βοηθούν να προχωρήσουμε όσον αφορά την την ε, πρόβλεψη ε, σε κάποιες πλημμύρες, σε κάποιες πάρα πολύ σχέσεις βροχοπτώσεις, ε, ο χρονισμός τους και έτσι μπορούμε να προτείνουμε καλύτερα τον κόσμο. Μπορούμε επίση έτσι να υπολογίσουμε το, το, το κίνδυνο, τη διακινδύνευση όσον αφορά ε, τι διάφορε θεομηνίε εκτό από τι ε, πλημμύρε. Επομένω, έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία, καλύτερο συντονισμό μεταξύ τη Ευρωπαϊκή ε, πρωτοβουλία για το διάστημα και των πρωτοβουλειών των αντιστοίχων των κρατών μελών. Ο τρίτο άξονα για να περιστρέφεται αυτή η υπόθεση, αυτό το πρόγραμμα είναι οι υπηρεσίε. μπορούμε να εμπλέξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά την συλλογή δεδομένων, όσον αφορά την λήψη κάποιων ε, εικόνων, φωτογραφιών ε, και τον συσχετισμό τους. Και έτσι είναι δυνατόν να εξυπηρετούν ε, περισσότερες χώρες ταυτόχρονα. Επομένως, έτσι κάνουμε βήματα προς τα εμπρός, τα πρόοδο όσον αφορά την τεχνολογία και κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε κάπως αυτόνομοι όσον αφορά αυτά τα τόσο σημαντικά δεδομένα, αυτές τις τόσο σημαντικές πληροφορίες και δεν θα εξαρτώμεθα από άλλες χώρες με τις οποίες εξαρτώμεθα σήμερα για τη λήψη αυτών των δεδομένων. Επίσης, ε, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση, ούτω ώστε να υπάρξει η αναγκαία υποδομή που θα μπορέσει να υποστηρίξει με τα δεδομένα που χρειάζεται τις εφαρμογές ε, αυτού του, του, προγράμματος. Και... Ε, αυτό το θέμα θα συζητηθεί και άλλο σήμερα, δηλαδή η μείωση των εκπομπών. Να αντιμετωπίσουμε την απερίμεση των δασών και αυτό βεβαίως απαιτεί πιο άμεση γνώση, πιο ενδελεχή, λεπτομερή γνώση όσον αφορά ε, την, την κάλυψη της γης από τα δάση. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλύτερη διαχείριση, με μεγαλύτερη ακρίβεια όσον αφορά το τι χρειάζεται από πλευράς χρηματοδοτικής. Πρέπει να δώσουμε τα κράτη που κατέχουν αυτά τα δάση, ούτως ώστε να δοθούν κίνητρα για τη διατήρηση των δασών. Κίνητρα στα κράτη. Ούτως ώστε να θεωρηθούν και ως δεξαμενές δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και να υπάρξουν ε, οικολογικές υπηρεσίες ε, για να εξασφαλιστεί ε, ένα σωστό κλίμα και η βιοπικιλότητα. Αυτά τα πράγματα τα ενέταξα στο κείμενο, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε τους κατάλληλους πόρους για αυτές τις αντισταθμίσεις και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι πόροι στο εσωτερικό του συστήματος εμπορίας εκπομπών ε, την χάνουν πιο αυστηρής διαχείρισης. Τέλος, θα ήθελα να ξανατονίσω ότι όλα αυτά εντάσσονται στα διαστημικά προγράμματα και στο ΓΚΕΟΣ, ε, στο Παγκόσμιο ε, Σύστημα Γεωπαρατήρησης. Στο Παγκόσμιο Σύστημα Συστημάτων Γεωσκόπησης. Πρέπει να τονίσουμε ότι τον ε, Ιανουάριο, Δεκέμβριο-Ιανουάριο 2014 ε, μπορούν να γίνουν ψηφοφορίες για τα οικονομικά θέματα. Θα πρέπει να επιμείνουμε ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι πόροι. Γιατί τόσο για την κατασκευή των δορυφόρων όσο και για την εκκίνηση των δορυφόρων θα πρέπει να δεσμευτούμε εκ των προτέρων, δύο-τρία χρόνια νωρίτερα. Εάν γίνει αυτή η ψηφοφορία, υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσουν τα πράγματα πολύ και υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί το κόστος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε συνολικά ότι το, το πρόγραμμα GMES, το πρόγραμμα ε, για την, τα συστήματα, το σύστημα γεωσκόπησης μπορεί να προχωρήσει. Πιστεύω ότι η πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή. Προτείνω τέσσερις τροπολογίες. Η πρώτη τροπολογία αφορά την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και το μετριασμό της αύξησης θερμοκρασίας του κλίματος και όλα τα δεδομένα ε, με τα οποία μπορεί να βοηθήσει αυτό το πρόγραμμα για αυτά τα θέματα. Την αναφορά επίσης στο σύστημα ΓΕΟΣ και το, η τρίτη τροπολογία αφορά την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία της Κομπαϊχάγης που θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο αναφοράς. Εκεί θα πρέπει να συγκεντρώνονται τα δεδομένα. Πολύ χρήσιμα δεδομένα, έτοιμα δεδομένα και συγκρίσιμα δεδομένα θα, θα συγκεντρώνονται εκεί στην Κοπενχάγη. Η τελευταία τροπολογία αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότηση του GMES, με τα έσοδα της Mission, ε, α, Emission Trading System, του ETS δηλαδή. Το σύστημα μπορεί να δώσει πολύτιμα δεδομένα, πολύτιμα στοιχεία, τόσο για την κλιματική αλλαγή όσο και για την αύξηση θερμοκρασίας του πλανήτη. Και επίσης μπορεί να δούμε τι μπορεί να γίνει με τα χρήματα, με τις αποζημιώσεις δηλαδή που προέρχονται από το ETS. Σας ευχαριστώ πολύ. Βιτόριο Πρόντι. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Συμφωνώ οπωσδήποτε ένα θέμα που ιδιαίτερα την δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ενδιαφέρει, διότι είναι σχετικό με τους στόχους μας. Και πάντα το έβρισκα κρίμα ότι το GMES είναι μια περίπλοκη έννοια και από πλευρά ορολογίας δεν βρήκαμε κάτι πιο απλό. Έχουμε τον Γαλιλαίο, τον Έρασμο, τον Λεωνάντο Νταβίντσι τα ξέρουμε ποια είναι αυτά, αλλά GMS e τι είναι αυτό. Μόνο οι επαΐοντες γνωρίζουν τι είναι αυτό, οι ειδικοί. Και ακούσαμε πόσες εφαρμογές υπάρχουν. Η παρακολούθηση της ε, καύσης ε, των δασών για αποψήλωση με δασοπυρκαγιές όλες αυτές ε, οι υποθέσεις των πλημμυρών, καταιγίδων για τις κλιματικές αυτές τα κλιματικά φαινόμενα πρέπει να ενδιαφερθεί η δική μας Επιτροπή. Είναι μια σημαντική έκθεση. Δεν πρέπει μόνο τεχνικά να την αντιμετωπίζουμε και πολιτικά έχει μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ για την παρουσίαση της έκθεσης. Έχουμε τον κύριο Ταπταρέλα που ζήτησε τον λόγο. Ο Σαλβατόρε από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Πρόντι εξέφρασε μια θετική γνώμη για αυτό το πρόγραμμα. Συμμερίζομαι απόλυτα αυτή τη στάση και αυτή τη γνώμη του. Και ευχαριστώ τον εισηγητή που με κάλεσε στη συνεδρίαση που είχαμε με τον διευθυντή του GMES που μας επέτρεψε να εμβαθύνουμε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Συμφωνώ με όλα όσα αναφέρει η έκθεση Πρόντι. Υπάρχει ένα μοναδικό στοιχείο για το οποίο κρατάω μία επιφύλαξη. Θέλω, θα ήθελα να το μελετήσω. Και αυτό είναι η σχέση μεταξύ αυτού του προγράμματος και του συστήματος ETS, ε, εμπορίας των εκπομπών δηλαδή. Καταλαβαίνω την άποψη του κυρίου Πρόντι. Νομίζω ότι εκείνο θέλει να βρει επιπλέον κονδύλια για τη χρηματοδότηση. Αλλά όμως ε, σε τεχνικό και νομικό επίπεδο θα πρέπει να δούμε αν αυτό που λέει είναι εφικτό. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη αναφορά, ρητή αναφορά και στο πρόγραμμα ΓΕΟΣ. Θα περιοριστώ σε αυτή τη σύντομη παρέμβαση να, εξηγήσω για να θέσω δύο ερωτήσεις προς την Κομισιόν και για να εκφράσω φυσικά μια θετική συνολική γνώμη. Ε, ο κ. Πρόεδρε είπε πάρα πολλά ε, θετικά στοιχεία, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα σημαίνει ότι εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτούμε μια σειρά δεδομένα πάρα πολύ σημαντικά και τα, τα παίρνουμε από οποιαδήποτε από και αφορούν αυτά τα δεδομένα οποιοδήποτε τμήμα του πλανήτη. Ε, τα έχουμε 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Ε, είτε ο ουρανός είναι νεφοσκεπής, είτε είναι ανεφέλωτος. Ε, και έτσι έχουμε στοιχεία για το περιβάλλον, αλλά και στοιχεία για την ασφάλεια. Μιλάω για πλημμύρες, καταολιστήσεις, χιονοστιβάδες, όλα όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε από καιρού καιρών. Επομένω, αυτό το σύστημα και αυτό το πρόγραμμα ε, είναι ένα δορυφορικό πρόγραμμα που ονομάζονται φρουροί. Είναι πέντε φρουροί που τοποθετούμε στο διάστημα και που μας δίνουν ε, μία σειρά από δεδομένα πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, υπόθηκε και τον κύριο Πρόντι, ότι μπορούμε παραδείγματο χάρη να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να προλάβουμε τι ε, πυρκαγιέ, όπω συνέβη πρόσφατα στην Ελλάδα. Ε, αυτοί οι δορυφόροι μα δίνουν τέτοια δεδομένα. Μπορούμε να, να προλάβουμε τι ε, προ... πυρκαγιέ. Επίση, ε, μπορούμε να εμποδίσουμε τη ρήπανση των ποταμών από τη βιομηχανία, το επίπεδο των νερών. Ακόμη και για τη θάλασσα είναι χρήσιμο. Παραδείγματο χάρη στην Κίνα υπήρχε ένα πρόβλημα με τα φύκια. Θα πρέπει να μπορούμε να δούμε πώς αναπτύσσονται αυτά τα φύκια και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα αφαιρέσουμε από τις θάλασσες. Μία σειρά από δεδομένα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χάρη σε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα επίσης, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, ε, σημαίνει και έρευνα και τεχνολογία και απασχόληση για τις επιχειρήσεις μας και τις βιομηχανίες μας. Επίσης, σημαίνει εξασφάλιση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια τεράστια πρόκληση, πολύ σημαντική και αυτό είναι ένα από αυτά τα προγράμματα που η κοινή γνώμη θα τα περάσει λίγο στον Τούκου. Δεν, θα τα, δεν τα γνωρίζει. Ε, όπως είπε και ο πρόεδρος, είναι τεχνική όρη αυτή και ο κόσμος δεν τους ξέρει. Όμως είναι ένα από αυτά τα προγράμματα που είναι απίστευτα χρήσιμη για όλους τους ε, πολίτες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ας πάω στις δύο ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Διάβασα κάπου που γράφτηκε για αυτό το πρόγραμμα, ότι πολλοί, πολλές από τις υπηρεσίες παρατήρησης της γης, της γεωσκόπησης, στην Ευρώπη δεν είναι αξιόπιστες, γιατί έχουν ε, διαρθρωτικές ελλείψεις. Και επίσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία μακροπρόθεσμα. Αυτό το στοιχείο το ανέφερε επίσης ο κύριος Πρόντιο. Το θέμα του, του μακρού χρονικού ορίζοντα. Και εδώ θέτω το πρόβλημα των χρηματοδοτήσεων. Εμείς έχουμε προγραμματίσει τις χρηματοδοτήσεις μέχρι το 2014. Υπάρχει και το θέμα της κατασκευής, ε, των, για την κατασκευή μάλλον των δορυφόρων. Και εν συνεχεία θα πρέπει να τους θέσουμε σε τροχιά 2014-2017. Αυτή η περίοδος 2014-2017 ε, είναι πολύ σημαντική για την εκτέλεση του προγράμματος και δεν έχουν προβλεφθεί χρηματοδοτήσεις. Σήμερα θα πρέπει να το θέσουμε αυτό το πρόβλημα. Ε, γιατί πρέπει να προβλέψουμε αρκετά εγκαίρως. Ε, για να, θέσουμε, να αποφασίσουμε θα θέσουμε σε τροχιά τους δορυφόρους πρέπει να το έχουμε προγραμματίσει δύο χρόνια πριν. Ε, επομένως πρέπει να προβλέψουμε πολύ νωρίτερα τις ε, χρηματοδοτήσεις. Γι' αυτό ακριβώς ο κ. Πρώτη προέβλεψε ότι ένα τμήμα των ε, κερδών από το ETS μπορούν να πάνε σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το κοινοβούλιο και αυτή η επιτροπή, η δική μας κοινοβουλευτική επιτροπή, θα πρέπει να εκκινήσει και να συντονίσει ένα διαθεσμικό διάλογο με τον πρόεδρο Μπαρόζο. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τον Μπαρόζο αν αυτό το πρόγραμμα είναι ένα από τα προγράμματα προτεραιότητας που έχει η Επιτροπή του. Σε, αυτό το διαθεσμικό πλαίσιο, φυσικά, θα πρέπει να εμπλέξουμε και την διαστημική υπηρεσία της Κοπενχάγης. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι το θέμα της governance γίνεται και περιβαλλοντικό θέμα, θέμα διαχείρισης των δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θέση έχει απέναντι στις ε, εθνικές ε, υπηρεσίες. Ε, για το θέμα της διαχείρισης των δεδομένων. Πώς διαφρώνονται όλα αυτά μεταξύ τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ταταρέλα. Βλέπω αυξάνεται ο ενθουσιασμός για το GNS και δίκαια. Τρίτος ο κύριος Ορεστερόση. Φαίνεται είναι ιταλικό επίπεδο αυτή η συζήτηση. Παρακαλώ. <laughs> Ε, πρόεδρε, ίσως γιατί ο εισηγητής είναι Ιταλός. Ε, μας ε, δίνει έτσι ενθουσιασμό αυτό και μας δίνει την όρεξη να κάνουμε ερωτήσεις. Ο, με τον σύντροφο κύριο Πρόντι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωπαρατήρησης, γιατί συχνά συνειδητοποιούμε ότι οι φυσικές καταστροφές, αν τις παρατηρήσουμε έγκαιρα, θα μπορούσαμε να τις αποφύγουμε, ή εν να τις αντιμετωπίσουμε. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρώπη να προγραμματίσει και να χρηματοδοτήσει μια τέτοια δομή, ένα τέτοιο, μια τέτοια υπηρεσία που θα παρατηρεί τους ωκεανούς, τις κλιματικές αλλαγές, τα ευαίσθητα δεδομένα για τη γη. Μην ξεχνάμε ε, τα προβλήματα της μόλυνσης ε, ή τα προβλήματα που αφορούν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και τις κλιματικές αλλαγές. Για όλα αυτά θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό το πρόγραμμα. Ε, γιατί έχουμε όμως κάποιες αμφιβολίες. Επειδή και πολλά κράτη, όπως η Ιταλία, Φερρυπίν, σήμερα έχουν ε, μία δέσμοι δομών ε, που έχουν, παραδείγματο χάρη, την ε, στρατιωτική βάση αυτή από όπου παρατηρούμε την ε, Μεσογειακή Λεκάνη ή άλλες δομές για την παρατήρηση της Αδριατικής. Έχουμε άλλες υπηρεσίες που ασχολούνται με τα δάση, τους ποταμούς. Έχουμε διάφορους φορείς δηλαδή. Έχουμε ένα σύνολο φορέων δικτυωμένων που ελέγχουν την επικράτειά μας. Φυσικά έχουν περιορισμούς. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έτσι μια σφαιρική θεώρηση. Το ερώτημα μου ποιο είναι. Όλοι αυτοί οι μικροί φορείς που όμως ε, προκαλούν και επισύρουν δαπάνες για τα κράτη-μέλη. Πώς θα καταλήξουν. Θα υποστηρίξουν αυτό το νέο φορέα, αυτό το νέο σύστημα, αυτή τη νέα δομή ή θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα και επομένως θα έχουμε μικροεπικαλύψεις, περιτές προφανώς. Αυτό το νέο πρόγραμμα, αυτό το νέο σύστημα που θα είναι και ένας οργανισμός που θα ελέγχει και την ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς ε, και την, και την ασφάλεια επίσης. Θα δίνει σε real time α, πληροφορίες στα κράτη-μέλη. Και επομένως ε, θα υπάρξει μια γενική εξοικονόμηση για πράγματα που κάποτε κάνανε άλλοι φορείς όπως αυτή που σας ανέφερα σε εθνικό επίπεδο και σε υποεθνικό επίπεδο τώρα για το ETS. Νομίζω ότι θα ήταν επικίνδυνο να χρησιμοποιήσουμε χρηματοδοτήσεις από το ETS. Ε, φοβόμαστε ε, όλο, γενικά το, το σύστημα της, του ETS ε, μπορεί, μπορεί, να εξοκύλει ε, με περίεργα παράγωγα στο μέλλον κτλ. Φοβόμαστε ότι για το θέμα της ε, κλιματικής αλλαγής το GMES ε, μπορεί να ε, γυρίσει μπούμεραγκ. Επομένως, οι ερωτήσεις μας είναι αυτό το GMES θα αντικαταστήσει όλους αυτούς τους μικρούς φορείς που κάθε κράτος, κάθε περιφέρεια της Ευρώπης έχει. θα έχει σταθερή σχέση με αυτούς τους φορείς και με τα κράτη-μέλη. Και Τι θα γίνει ε, με τη χρηματοδότηση από τις ποσοστώσεις ε, του ETS, ε, τις εποστώσεις και τις εκπομπές στα πλαίσια του ETS. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. δεν είναι μόνο οι Ιταλοί που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόντι για την έκθεσή του. Το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μοιάζει τεχνικό, αλλά είναι και εξόχως πολιτικό. το να έχουμε ακατέργαστα δεδομένα. Γιατί περί αυτού πρόκειται τελικά, έτσι. Από τη μία, μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τις δημόσιες πολιτικές. Γιατί ο κόσμος λέει πολλά. Πολλοί λένε πολλά. Το θέμα είναι τι συμβαίνει. Ε, πώς αποτελεσματικοί είμαστε με τα συστήματά μας και τις πολιτικές μας. Θα, αποκτήσουμε λοιπόν ένα εργαλείο που θα μας επιτρέψει να πάμε πέρα από τους εθνικούς ελέγχους. Πέρα από την ε, θαυμάσια δουλειά που κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος ε, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των δεδομένων. Θα έχουμε στοιχεία ενημερωτικά με πολύ πιο προσπελάσιμο τρόπο, παραδείγματο χάρη για τις θάλασσες. Για τις θάλασσες ήταν δύσκολο να έχουμε στοιχεία, γιατί είμαστε στο τομέα της εξοεδαφικότητας. Επομένως αυτό το στοιχείο είναι εξόχως ε, σημαντικό. Επίσης είναι και ένα δημοκρατικό εργαλείο. Αν θέλουμε τις δημόσιες πολιτικές αυτές να τις αναπτύξουμε, αν θέλουμε οι πολίτες μας να είναι θετικοί απέναντι στις πολιτικές πρόθεσης και προστασίας βιοποικιλότητας θα πρέπει να ενημερώνονται σωστά. Και αυτά τα στοιχεία που θα μας δίνει αυτό το σύστημα ε, θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους να παρακολουθούν τις εξελίξεις ε, και τα τεκτενόμενα. Θα τους επιτρέψει να είναι πολύ πιο απαιτητικοί σε περίπτωση που οι πολιτικές που δημιουργούμε δεν αρκούν για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Τελευταίο σημείο. Ε, είναι δύσκολο να το συνδέσουμε αυτό με το κλίμα και καταλαβαίνω τις ε, προθυμίες που ακούγονται για τη σχέση του ενός με το άλλο. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή η διασύνδεση θα γίνει αναπόφευκτα. Δεν θέλω να πω ότι πρέπει να γίνεται και καλά σήμερα, γιατί ίσως είναι πολύ νωρίς και αντιπαραγωγικό ενδεχομένως, αλλά νομίζω ότι κάπου στο, βάθο βάθος του μυαλού μας θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτό το σύστημα που δημιουργούμε κάποια στιγμή θα μπορούσε να συνδεθεί με τις κλιματικές ε, αλλαγές μόνο και μόνο αν θέλετε και μόνο και μόνο για να ελέγξουμε τις κλιματικές αλλαγές αυτό. Και μόνο αυτό να κάναμε θα άξιζε αυτό το... Ζητώ συγγνώμη ε, που φτάνω αργά. Νομίζω ότι διάφορες συχνότητες έχουν δοθεί σε αυτό το πρόγραμμα για να επιτραπεί η διάδοση των ε, πληροφοριών. Θα γίνουν σεβαστές αυτές οι συχνότητες. Ε, για το Γαλιλαίο, με βάση πληροφορίε, υπάρχουν κάποιε ανησυχίε ε, για την κινέζικη επικράτη, όπου οι συχνότητε δεν έχουν γίνει σεβαστέ από του Κινέζου. Ε, Συνήθω αυτέ οι συμφωνίε είναι συμφωνίε κυρίων. Πώ σκοπεύετε να διατηρήσετε τι ε, συχνότητε, αν έχουν ήδη δοθεί συχνότητε για αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε. Δεν βρέπω να ζητούν άλλοι τον λόγο. Μου λένε, μαθαίνω ότι το πρόγραμμα Είχε το όνομα Κοπέρνικος παλαιότερα, αλλά κάποιος είχε αυτό το όνομα δικαιόχρηση με αυτό το όνομα και έτσι υπήρξαν νομικές δυσκολίες. Υπάρχουν και άλλες ίσως ιδέες. Να το προτείνουμε. Να υπάρχει, ας το πω έτσι, μία ε, ταύτιση ώστε να ξέρει ο κόσμος τι είναι το GVS. Ο κύριος Μουτατιέ παρακαλώ από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλές ερωτήσεις ακούσατε, παρακαλώ απαντήστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύει η Επιτροπή σας ε, για την πρότασή μας που είναι πρόταση που θα αφορά αυτό το πρόγραμμα παρατήρησης της γης που εκπονήσαμε για να απαντήσω ε, όσον αφορά τη διασύνδεση των δραστηριοτήτων που θεωρούμε ότι θα αποτελούν μια προστιθέμενη αξία ε, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες ε, κινήσεις που έχουν γίνει από κράτη-μέλη, το οποία θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Γιατί το GMS, το GMS ακριβώς έτσι συνελήφθη, ακριβώς έτσι ε, τον εμπνεύτησαν επί τη βάση των δραστηριοτήτων των κρατών μελών. Και υπάρχει και αυτός ο άξονας που αφορά το διάστημα που είχε ως αφετηρία μία ανάλυση. Μία ανάλυση που θα έπρεπε σε ενωσιακό επίπεδο να συμπληρωθεί. Επομένως, το GMES δεν πρόκειται να αναστείλει τα προγράμματα των κρατών μελών, ούτε πρόκειται να παραβλάψει κάποιες αναδυόμενες αγορές όσον αφορά για την ε, ε, διάχυση αυτών των πληροφοριών. Τώρα, όσον αφορά την εντολή προς τις αρχές που χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες στα κράτη-μέλη, πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό, αναφέρθηκαν στην πολιτική προστασία, που είναι αρμοδιότητα διαφόρων αρχών στα κράτη-μέλη. Βεβαίω και παραμένει το GMS πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και καταρχήν είναι ένα εργαλείο. Με ένα τέτοιο εργαλείο δεν πρόκειται να θέσουμε σε αμφισβήτηση την, ε, τις αρμοδιότητες, την εντολή των διαφόρων αρχών και φορέων στην Ευρώπη που έχουν για δουλειά τους να προστατεύσουν τους πολίτες. Άρα θα υπάρξει κάποια ε, αμοιβαία εκμετάλλευση κάποιων ε, ε, έργων υποδομής, τόσο ώστε οι διάφοροι χρήστες των κρατών μελών να ωφεληθούν στο έργο τους. Τώρα για την χρηματοδότηση, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα χρηματοδότησης που να μπορέσει να μας ε, αποδώσει όσο γίνεται περισσότερο στον αυτό και την ωφέλεια. Σας παραπέμπω στην ανακοίνωσή μας όσον αφορά την ε, διάσταση που αφορά το διάστημα, τη διάσταση του GMS που αφορά το διάστημα, διότι έχουμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε κάποιες προκλήσεις και θα πρέπει να ληφθούν μέχρι το 2011 συγκεκριμένες αποφάσεις ούτως ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο το GMS μέχρι το 2011. Επίσης, λέει η να μας ότι για μια σειρά παρατηρήσεων που σήμερα γίνονται από τα κρατη θα συνεχίσει η συνεργασία, η αρρωγή προς τα κρατη και θα υπάρξει ένα σχήμα εταιρική σχέσης για το μέλλον μεταξύ κρατών μελών και ένωσης. Τέλος, όσον αφορά τη συχνότητα ή τις συχνότητες, δεν είναι πρόβλημα σήμερα όσον αφορά το GMS. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα vielen Dank. ευχαριστώ πολύ για την χρηματοδότηση μεταξύ 2014-2017, θέμα που ανέφερε ο κύριος Ταταρέλα, υπάρχει ένα κενό εκεί. Τι θα γίνει, τι φαντάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση αυτή. Oui, donc en, ce qui concerne les, les financements qui devraient être inscrits, donc les disponibilités Να δούμε τι κονδύλα θα πρέπει να στον ε, για το 2017. Αυτό θα ενταχθεί βεβαίως στην διαδικασία της χάραξης της δημοσιονομικής πολιτικής και του χρηματοοικονομικού πλαίσιου που θα κινηθούμε για τον προϋπολογισμό και από τον Οκτώβριο άρχισε να λαμβάνονται κάποιες ε, αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν και άλλες όσον αφορά τις δραστηριότητες που θα πρέπει να αναλάβουμε για αυτό το, το διάστημα 2014-2017 και να υπάρχει βέβαια ε, αναγκαία ε, κάλυψη και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε απαρακόλλητη δραστηριότητα και χωρίς διακοπές όσον αφορά την παρατήρηση του διαστήματος. Κατά αυτόν τον τρόπο είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε τις μονάδες Β να υπάρχει να υπάρχουν τα κατάλληλα έργα υποδομή όσον αφορά επίσης εκτόξευση δορυφόρων και καθ' τον τρόπο να υπάρχει η κατάλληλη δημοσιονομική στρατηγική και μέχρι το 2011 αυτή να έχει εκπονηθεί και ολοκληρωθεί στα πλαίσια του σημερινού δημοσιονομικού πλαίσιου ακόμα και αν αυτέ οι δραστηριότητε θα πρέπει να αρχίσουν να, τρέχουν, να αναπτύσσονται από το 2014. Βιτόριο Πρόντι για τις τελικές παρατηρήσεις παρακαλώ. Ε, io credo che sia stata una discussione molto interessante. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η φάση της συζήτησης. Ευχαριστώ κυρίως τον κύριο Ταταρέλα για την συνεισφορά του. Θα ήθελα να τονίσω ότι το σύστημα ανταλλαγής ε, εκπομπών, εμπορίας εκπομπών ε, με το GMES, ε, θα πρέπει, αυτά τα δύο συστήματα θα πρέπει να αρθωθούν με τρόπο συνεκτικό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την αύξηση θερμοκρασίας του πλανήτη και διάφορες δραστηριότητες γύρω από τις κλιματικές αλλαγές. Το ETS το θεωρώ λοιπόν σημαντικό εργαλείο. Και νομίζω ότι πραγματικά έχει νόημα να απαιτήσουμε το σύστημα ETS να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του GMES. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, όπως ε, πρότεινε η Επιτροπή ε, και στα πλαίσια της ε, διάσκεψης Κοπενχάγης. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτή την προοπτική του ETS, δηλαδή. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε επίσης κάποιες φορολογικές αλλαγές, ότι το βάρος από τα εισοδήματα θα πέσει τώρα ε, στη χρήση των φυσικών πόρων, δηλαδή σε αυτούς που χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους. Θα μετατεθεί το βάρος από τα εισοδήματα εκεί. Έχει νόημα αυτή η εξέλιξη. Και προς τα εκεί πηγαίνουν τα πράγματα. Ε, προς τον κύριο Ρώση θέλω να πω, ναι, είμαστε καλοί σύντροφοι. Σύντροφοι πορείας. Και νομίζω ότι οι δορυφόροι μπορεί να μας βοηθήσουν για να βρούμε τη σωστή πορεία. Και πιστεύω ότι ο κύριος Ρώση θα το μετανιώσει, αν συμφωνήσει μαζί μου. Επίσης, για τις δομές ελέγχου, τις οποίες αναφέρει το έγγραφο ως ε, επιτόπιες παρατηρήσεις. Αυτή είναι η συνιστόσα επιτόπιων παρατηρήσεων. Νομίζω ότι η επισκόπηση που κάνει το GMES και η επιτόπια επισκόπηση μπορούν να συνδεθούν. Εγώ θα μπορούσα να το ονομάσω Μάρκο Πόλο. Επισκόπηση Μάρκο Πόλο. Ε, Κάποιο άλλο βουλευτή λέει, γιατί όχι, εγώ θα μπορούσα να το ονομάσω Βιτόριο Πρόντι. Όχι, όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν θέλουμε να τροφήσουμε κάποια άτομα εδώ. Με τις νέες ε, επισκοπήσεις μπορούμε να έχουμε και μια σωστότερη χαρτογράφηση. Δηλαδή, ανάμεσα στα δορυφορικά δεδομένα και στα τοπικά δεδομένα μπορεί να υπάρξει μια διασύνθεση. Επίσης τα δεδομένα αυτά είναι συγκρίσιμα. Ακριβώς γι' αυτό έβαλα μία τροπολογία για την υπευθυνοποίηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, η οποία έχει την ευθύνη της οργάνωσης, θα μπορούσε να έχει την ευθύνη της οργάνωσης των δεδομένων των επιτόπιων. Επίσης, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε το GMES είναι ένα σύστημα για την ε, λεπτομερή παρατήρηση της κατάστασης του εδάφους. δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή η οδηγία για την προστασία του εδάφους. Πολύ σημαντική. Το GMES θα είναι ένα εργαλείο που θα μας επιτρέψει να έχουμε λεπτομερείς ε, παρατηρήσεις για το έδαφος, την βλάστηση, την ε, υγρασία του. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει και με αυτή την οδηγία για την προστασία του εδάφους. Υπάρχει μια αναντήρητη ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία. Εγώ πραγματικά περιμένω πολλά. Και ελπίζω τώρα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και με τις ε, χρηματοδοτήσεις. Ε, ελπίζω να μην γίνει ψηφοφορία αυτή για την οποία σας μίλησα πριν, γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Σε ευχαριστούμε συνάδελφε Πρόντι. Επί τη ουσία αρμόδια η επιτροπή είναι η Επιτροπή Ήτρε. Ο συνάδελφο Γκλάντ έχει να λάβει τη σύνταξη έκθεση δεν θα μπορεί να ονομάζεται πρώτη το πρόγραμμα, μια και ο Γκλάντια το έχει αναλάβει, αλλά Μάρκο Πόλο καλό όνομα Κάτι το οποίο θα μένει και θα το θυμάται ο πολίτης είναι το ευκταίο προθεσμία για τις τροπολογίες 17 Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι. Εντάξει. Περνάμε τώρα στο σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης. Ποιο είναι αυτό? Η αηφορία στο μέλλον των μεταφορών. Εδώ η Επιτροπή Μεταφορών η κύρια αρμόδια επί της ουσίας. Εμείς όμως σωστά αποφασίσαμε να συντάξουμε γνωμοδότηση την οποία ανέλαβα να συντάξω εγώ ο ίδιος. Έχουμε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ προπαρασκευάζεται μια νέα λευκή βίβλος για το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη. Το παλαιό διάστημα 2010 το 2010 εκπνέει η παλαιότερη θα έλεγα διάρκεια του προγράμματος και τώρα πρέπει να προβληματιστούμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι το 2020, πώς θα διοργανώσουμε τις μεταφορές πανευρωπαϊκά. Και πραγματικά πολλά θέματα εδώ αφορούν τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εγώ έχω οκτώ προτάσεις που υπέβαλα και που μπορούμε να καταθέσουμε όσον αφορά την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών που είναι αρμόδια επί της Πρώτον, να πούμε ότι δεν καταφέραμε ακόμα το εξωτερικό κόστος των μεταφορών να το εσωτερικεύσουμε όσον αφορά το κόστος ε, των μεταφορών, να υπολογιστεί εσωτερικά. Αυτή είναι η συζήτηση που πολλές δεκαετίες διεξάγεται. Δηλαδή, polluter pays, ο ρηπαίνων πληρώνει. Αυτή είναι η αρχή και πρέπει έτσι να καθορίζεται και να αντανακλάται στο εσωτερικό κόστος. Αυτό θα είχε επιπτώσεις στην επιλογή πιο φιλοπεριβαλλοντικών μέσων μεταφορών σε σχέση με τα λιγότερο φιλοπεριβαλλοντικά μέσα ε, οι μεταφορών. Μετά το πρόβλημα των πόλεων. Και εδώ πάλι ένα πρόβλημα μεταφορών και ε, κυκλοφορίας. Έχουμε αυτό το πρόβλημα των πόλεων. Χρειαζόμαστε για τις πόλεις και για το περιβάλλον τους και για τον υπαίθριο χώρο θελκτικά συστήματα μεταφορών που θα είναι φιλοπεριβαλλοντικά. Ακριβώς σε κέντρα με πυκνή δόμηση και κατοίκηση, στις πόλεις δηλαδή, στα αστικά κέντρα, βλέπουμε ότι η ποιότητα της ατμόσφαιρας του ατμοσφαιρικού αέρα είναι κακή και αυτό οδηγεί σε προβλήματα υγείας. Αυτό οδηγεί στην ιδέα ζωνών, ξεχωριστών ζωνών περιβάλλοντος, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να βελτιωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και να έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα όπου δεν θα μολύνεται. Ο θόρυβος είναι μάστιγα για εκατομμύρια ανθρώπους η όχληση από τον θόρυβο. Πρέπει να μπορέσουμε να μειώσουμε το επίπεδο της ε, ηχητικής όχλησης και παράλληλα με τις εκπομπές ρήπων διοξιδίου του άνθρακα που έχουν αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό Έχουμε και άλλες εκπομπές ρήπων, όπως ε, τα οξύδια του αζότου, το ε, θείο, τα, τα, το διοξίδιο του θείου και άλλες εκπομπές ρήπων που μέχρι το 2020 θα πρέπει να μειωθούν πολύ σε σημαντικό βαθμό. Στο σημείο 6 αναφέρω τις ναυτιλιακές μεταφορές που αυξάνονται και αυτές και πρέπει να συνεισφέρουν από πλευρά του ε, για την προστασία του περιβάλλοντο και την προστασία του κλίματο. Ε, οι ναυτιλιακές μεταφορέ ε, είχαν εξαιρεθεί μέχρι σήμερα από το σύστημα εκπομπών ρήπων και όπω λέμε και στην πρόταση ψηφίσματος για το κλίμα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι ναυτιλιακές μεταφορές όπως και οι αέριες μεταφορές με αεροπλάνα, πράγμα το οποίο έχουμε αποφασίσει και εγκρίνει. Μετά χρειαζόμαστε τεχνολογική καινοτομία ώστε να είναι πιο πράσινες οι μεταφορές στην Ευρώπη. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει διαφορετική ισορροπία. Όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία είναι ισχυρή, είναι πανίσχυρη, έχει πάμπολα κονδύλια και κάνει και έρευνες. Πάει όμως πολλές φορές στην λανθασμένη κατεύθυνση. Έχουμε όμως την ελπίδα ότι θα κατευθυνθεί προς την σωστή κατεύθυνση. Οι σιδηρόδρομοι όμως δεν έχουν πολλά κονδύλια και ούτε κάνουν έρευνες ε, σχετικά. Και τα αστικά κέντρα και οι μεταφορές είναι πολλές φορές ε, ελληματικές και δεν μπορεί κανείς να ε, χρησιμοποιήσει, δεν γίνεται από το κράτος ε, η επιδότηση όπως γίνεται πολλές φορές όσον αφορά την αυτοκίνητο βιομηχανία και αυτό είναι ένα θέμα των σιδηροδρόμων που θέλουμε να το προωθήσουμε Αυτά ουσιαστικά είναι από πλευρά μου θα έλεγα τα σημεία, τα κυριότερα σημεία που προτείνω για από πλευρά Επιτροπής Περιβάλλοντος για την Επιτροπή Μεταφορών. Έχουν ζητήσει συνάδελφοι τον λόγο τώρα. Χαιρετίζω βέβαια και μια ομάδα από την Αυστρία που με πρόσκληση της κυρίας Κάτερμπαχ έχει προσέλθει εδώ που ε, ενεργοποιούνται στα ευρωπαϊκά θέματα. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φίλοι μας χειροκρότημα. Ωραίο. Λοιπόν, ο Ματίας Γρότερ ζήτησε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Την νομοδότηση αυτή τη θεωρώ πολύ σημαντική. Το θέμα της πολιτικής μεταφορών σε τακτά διαστήματα το εγγράφουμε στην ημερήσια διάταξη και όσον αφορά τις ευρωπροδιαγραφές, δηλαδή όσον αφορά τις μειώσεις, ε, έχουμε εμεί συνεισφέρει με θετικό τρόπο μέχρι το 2014 με το Ευρω 5 για την ε, νομοθεσία για τις εκπομπές τρύπων και θα έχουμε και στη συνέχεια την Ευρω 6 για μικρά οχήματα. Βρίσκω ότι ο τομέα των βιοκαυσίμων και των εναέριων μεταφορών, σε αυτά τα δύο θέματα θέλω να αναφερθώ, θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία στη γνωμοδότησή μας. Οι σενέριες μεταφορές ένα σύστημα νομοθετικής διαβούλευσης για τις εκπομπές ρήπων είχε επιλεγεί. Ένα συμβιβασμός με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η τωρινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τη μείωση διοξιδίων του αζότου. Μας το υποσχέθηκαν αυτό και μέχρι σήμερα όμως δεν έγινε τίποτα, δεν υπέβαλαν σχετική πρόταση. Πιστεύω ότι στην έκθεση αλλά και εκ νέου ως Επιτροπή Περιβάλλοντος θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση, να ενεργοποιηθούμε ώστε να υποβάλουν αυτές τις προτάσεις το αργότερο με την νέα ε, ε, Επιτροπή που θα αναλάβει τις ε, τα χαρτοφυλάκια αυτά. Θέλουμε η υπόσχεση αυτή να τηρηθεί. Όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, εδώ νομοθετική δράση είχαμε το προηγούμενο έτος όσον αφορά και τα ανανεώσιμα και τα βιοκαύσιμα. Πρέπει να πάμε πιο πέρα όμως, να σκεφτούμε ακόμα πιο πολύ για να δούμε τι θα γίνει. Δεν πρέπει να δούμε κοντόθωρα τα πράγματα πολλοί ευρωβουλευτές είπαν η βιομάζα να χρησιμοποιείται εκεί που είναι πιο αποτελεσματική. Όμως πρέπει να ανοίξει η συζήτηση, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Η γνωμοδότηση εδώ θα μπορούσε να είναι το σωστό μέρος για να υποβάλουμε κάποιες προτάσεις. Πού μπορούμε να υποκαταστήσουμε κάτι. Δεν μπορούμε την κυροζήνη να την υποκαταστήσουμε. Χρειαζόμαστε όμως βιοκαύσιμα δεύτερης γενεάς εδώ, αλλά και σε άλλους τομείς και σε μεγάλες αποστάσεις εδώ μόνο τα βιοκαύσιμα μπορούν να βοηθήσουν και να δώσουν μια διέξοδο και οι μεγάλες, μεγάλων αποστάσεων μεταφορές ε, να μπορέσουν να, ε, να τα χρησιμοποιούν τα βιοκάσιμα. Θα επιθυμούσα να το κάνουμε αυτό σε αυτή τη γνωμοδότηση. Τώρα, το ευρωαυτοκόλλητο είναι ένα σημαντικό νομοθετικό ε, πλαίσιο. Το Κοινοβούλιο είπε ότι είναι υπέρ της Ευρωβινιέτας η Σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου, αλλά από ό,τι φαίνεται και η Ισπανική Προεδρία στη συνέχεια, αυτό το θέμα δεν θέλουν να το ε, προαγαγούν. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα σημαντικό πολιτικό μέσο, μέτρο, ώστε ε, η επόμενη, Προεδρία του Συμβουλίου να πάρει την σκητάλη και να αναλάβει πρωτοβουλίες. Το Συμβούλιο πρέπει να δραστηριοποιηθεί οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ματίας Γκρότε, ο Ρίχαρτ Ζέιμπερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα τον Ματίας Γκρότε, ιδιαίτερα στα όσα είπε, να τον υποστηρίξω, ιδιαίτερα στι τελικέ του παρατηρήσεις και για την Ευρωβινιέτα που επιτέλους θα πρέπει από πλευράς του Συμβουλίου να προωθηθεί και είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκείνο το οποίο έκανε πολλά πράγματα και η Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι με αυτόν τον τρόπο αποφασίσαμε να λειτουργήσει η Ευρωβινιέτα όπως έχει προταθεί. Δυστυχώς το Συμβούλιο δεν είναι πρόθυμο να αναλάβει τα αναγκαία μέτρα για να αρχίσει να ισχύει αυτό. Προέρχομαι από ένα ομοσπονδιακό κρατήδιο στην Αυστρία όπου έχουμε πολλά βαριά οχήματα, μεγάλα φορτηγά που περνούν από την περιοχή μας. Είναι πολύ σημαντικό η συμφόρηση των μεταφορών και της κυκλοφορίας ε, να βελτιωθεί όσον αφορά τους πολίτες μας. Στην έκθεση λέτε ότι θα πρέπει να εσωτερικευθεί το εξωτερικό κόστος στι μεταφορές και η Ευρωβινιέτα είναι ένα τέτοιο μέτρο. Μπορούμε να, πετύχουμε μέρος αυτού του στόχου με αυτό το μέσο. Και στην Αυστρία με αυτόν τον τρόπο έχουν συνεισφέρει ώστε να πετύχει αυτό. Αλλά τα κράτη-μέλη πρέπει επιτέλους να υπομισθούν τις ευθύνες τους, να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη και να υλοποιηθεί αυτό από πλευράς του Συμβουλίου. Δεύτερον, για την έκθεσή σας. Πολύ καλή είναι η έκθεσή σας και ζητώ πάλι η Ευρωβινιέτα ως θέμα να ενταχθεί και να προαχθεί πρέπει από πλευράς, ε, ε, την, μας τα ευχολόγια με την πραγματικότητα να τα διαχωρίζουμε. Αυξάνονται οι όγκοι μεταφορών και θα πρέπει να δούμε και την συμπεριφορά κινητικότητας ε, από πλευράς των πολιτών μας, πώς αλλάζει και πώς επηρεάζεται από πλευρά των πολιτικών μας πρέπει να βρούμε τις παραμέτρους ώστε η κινητικότητα αυτή να διαμορφωθεί σε σωστά πλαίσια. Να δώσουμε τα μέσα ώστε να είμαστε φιλοπεριβαλλοντικοί από τους φορεί μεταφορών που θα χρησιμοποιούμε επίσης ε, και την ε, μαζική μεταφορά και την ατομική μεταφορά με τα ταχύ. Το σημείο 7 έχει νομίζω κέρια σημασία, γιατί εδώ μπορεί να δώσουμε τις κατευθυντήρες γραμμές στους προσανατολισμούς, να μην κατηγορούνται οι πολίτες όταν χρησιμοποιούν το ταχύ τους ε, διαρκώς και αν δεν το καταφέρνουμε από πλευρά πολιτική να δημιουργήσουμε συνθήκε πλαίσιο ώστε να κατευθυνθούμε στη σωστή κατεύθυνση, οι πολίτε δεν ευθύνονται γι' αυτό. Δεν είναι εκείνοι που πρέπει να πληρώσουν τα σπασμένα επειδή χρησιμοποιούν το ΙΟΤΑΧ του, ελήψη άλλων πολιτικών και ατομικά χρησιμοποιούν το ΙΟΤΑΧ. Λοιπόν, εναέριε και θαλάσσιε μεταφορέ πρέπει να ενταχθούν. Δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση το πρόσχημα ότι είναι δύσκολο να υλοποιηθεί αυτό ο στόχο. Ε, που έχουμε ακούσει και στην Ευρωβουλή δεν μπορεί να είναι ε, αξιόπιστο. Πρέπει να ενταχθούν και οι ε, ναυτιλιακές μεταφορές στο σύστημα εκπομπών ρήπων και οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να υπομισθούν τις ευθύνες τους, να έρθουν στο ύψος των ευθυνών τους οι διεθνείς συμβάσεις να συναυθούν και να μπορέσουν να καλύψουν αυτή την ανάγκη των ναυτιλιακών μεταφορών. Λείπει η πολιτική βούληση. Αν υπάρξει μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει να το εντάξουμε στην έκθεση και να υπάρξουν οι κανονισμοί, οι διατάξεις εκείνοι. Σας εύχομαι συγχαρητήρια για την έκθεση έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε Ζέβε, Ο κύριος Τρεμόπουλος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι οι προτάσεις του εισηγητή ε, κινούνται σε μια σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να προσθέσω ε, κάποια σημεία. Όσον αφορά την ε, εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους των ε, μεταφορών, είναι μια πάρα πολύ σωστή ιδέα που έχουμε υπερασπίσει και σε αυτή την αίθουσα επανειλημμένα. Ε, πρέπει να συνοπολογίσουμε όμως σε αυτή την εσωτερήκευση και την απώλεια της βιοπικιλότητας αλλά και άλλα κοινωνικά κόστη, ιδιαίτερα ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας ε, που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Τα έσοδα της ε, εσωτερήκευσης του κόστους θα πρέπει να ε, δρομολογηθούν σε βιώσιμους τύπους μεταφορών και θα πρέπει να συνδυαστούν και με μέτρα προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές. Στην, στο σημείο 2 αναφέρεται η αυξανόμενη σημασία που έχει η χωροταξία για το θέμα που συζητούμε. Ε, θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο σαφές και να μιλήσουμε για ενίσχυση της αποκέντρωσης των λειτουργιών των πόλεων. Ε, επίσης, ε, μιλά για ελκυστικά συστήματα μαζικών ε, μεταφορών, όπου θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα, να αναφερθούμε ιδιαίτερα στα μέσα σταθερής τροχιάς ε, στο μετρό, στις μεγάλες πόλεις και στο τραμ. Ε, επίσης, ε, στο σημείο 3 αναφέρεται σε μέτρα εξομάλυνσης της κυκλοφορίας οχημάτων. Θα προτιμούσαμε την αλλαγή της λέξης σε αποθάρρυνση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, όπως πολύ σωστά είπατε και πριν, για το κέντρο των πόλεων. Ε, βεβαίως χρειάζεται μια μεγαλύτερη έμφαση στα κίνητρα για το περπάτημα και τη χρήση των ποδηλάτων. Ε, αυτό που πρέπει να τονίσουμε και να ζητήσουμε είναι να αποτελέσουν οι στόχοι της χάρτας των Βρυξελών για το ποδήλατο να αποτελέσουν τμήμα η, της επίσημης ευρωπαϊκής πολιτικής και της νομο, αντίστοιχης νομοθεσίας το Velocity Project πρέπει να χρηματοδοτηθεί παραπέρα, να ενταχθεί στο TEN-T δίκτυο, το οποίο πρέπει να εξυγχρονίσουμε και να αναθεωρηθεί με έμφαση σε πιο βιώσιμες μορφές ε, μεταφορών. Ε, θα ήθελα να προσθέσω ότι στο σημείο που αναφέρεται για ζώνες περιορισμένων εκπομπών θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και την πρόταση για ρυθμίσεις για χαμηλά επίπεδα ταχύτητας στα αστικά κέντρα. Ε, στο σημείο 5 ε, αναφέρεται ότι ε, οι οδικές μεταφορές έχουν περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές σωματιδίων PM10. Ε, α, αυτό ε, δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχουν περιορίσει σε κάποιες χώρες. Ε, στο, η έμφαση για την, ε, στο ίδιο σημείο για τη σταδιακή μετάβαση της μεταφοράς φορτίων από τις οδούς προς το σιδηροδρομικό ε, δίκτυο είναι κάτι πολύ σημαντικό θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια παραπάνω. Δεν θέλω να καταχραστώ άλλο το χρόνο. Ε, θα πω επίσης για το σημείο 7 ε, όταν αναφέρεται στον ρόλο της ε, τεχνολογίας λέει ότι μόνο μια ριζική αλλαγή στην τεχνολογία μπορεί να φέρει τη μείωση εκπομπών. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ μπορεί να φύγει η λέξη μόνο γιατί υπάρχουν και πολιτικές διαστάσεις όπως η αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης και δεν μπορούμε να αποθέσουμε τις, ε, τις ελπίδες μας μόνο στην τεχνολογία. Θα ήθελα να κλείσω με δύο επιπλέον ε, σημεία. Ε, το ένα αφορά την έμφαση και την αναφορά στην πρόσβαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, η οποία πρέπει να είναι ένα οριζόντιο στοιχείο στον σχεδιασμό των μεταφορών. Να αφορά δηλαδή όλα τα είδη μεταφορών. Και τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η συντήρηση ε, και η αναβάθμιση των υπαρχόντων υποδομών μεταφορών πρέπει να προηγηθεί της κατασκευής καινούριων υποδομών. Η επιδότηση καινούριων υποδομών πρέπει να εστιάσει σε φιλικά προς το περιβάλλον έργα, όπως οι δημόσιες μεταφορές, το τρένο, οι ποδηλατόδρομοι, οι συνδυασμένες μεταφορές και η οδική ασφάλεια γενικά νομίζω ότι μπορεί να είναι μια καλή βάση για να συνεισφέρουμε και εμείς σε αυτή τη συζήτηση και την πρωτοβουλία που παίρνετε. Πολύ σας ευχαριστούμε συνάδελφε Τρεμόπουλε. Η κυρία Ντεμπρόιν παρακαλώ. Ευχαριστώ, uh, Θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για τη δουλειά που κάνατε. Θα ήθελα να τονίσω, όπως κάνετε και εσείς, ότι ε, η παράγραφος 7 για την έρευνα και την ανάπτυξη είναι κεντρική σημασία. Το τόνισαν και άλλοι συνάδελφοι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με την ε, πρόταση του κυρίου Τρεμόπουλου για αυτή τη διαγραφή που πρότεινε. Δεν νομίζω θα χάσει τίποτα η παράγραφος. Δύο σημεία θα ήθελα να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε. Στην παράγραφο 2, μετά την παράγραφο 2, εκεί που μιλάτε για τις αστικές μεταφορές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι καλές δημόσιες διαφορές ε, συνδέονται με τις υπηρεσίες ε, στις περιοχές υπαίθρου και αυτό μας βοηθάει να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων από τα αυτοκίνητα. Στην τελευταία παράγραφο επίσης, εκεί που μιλάτε για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την πρωτοβουλία Σιβήτας, συμφωνώ με αυτά που λέτε εδώ, διερωτώ με απλώς αν μπορούμε να συμπεριλάβουμε και το κοντσέρτο, παρότι ασχολείται κυρίως με την ενέργεια. Αλλά χάρη σε αυτή την χαμηλή εκπομπή διοξιδίων του άνθρακα νομίζω θα μπορούσε να είναι τμήμα αυτού που αναφέρεται στο σημείο 8. Ευχαριστώ. Ωραίστε Ρώση, παρακαλώ. Είναι ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Παρότι συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που είπε ο κύριος Πρόντι προηγουμένως, είμαι σχεδόν ε, σύμφωνο και με αυτά που είπατε κι εσεί. Μόνο δύο υποσημειώσει. Να μην ξεχνάμε ότι η μόλυνση δεν συνδέεται κυρίω με τι μεταφορέ, αλλά με τι μολύνσει από τι κατοικίε. Ε, μην ξεχνάμε ότι και οι κατοικίε στα νοικοκυριά είναι πολύ σημαντικέ πηγέ μεταφορέ. Τουλάχιστον εξίσου με τι μεταφορέ. Επομένω, προσοχία. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις νέες μορφές θέρμανσης να μην τις ξεχνάμε αυτές. Το πρόβλημα λοιπόν της αύξησης θερμοκρασίας ε, του πλανήτη ε, οφείλεται στις μεταφορές αλλά και στα νοικοκυριά. Ε, λέτε πολλά ωραία πράγματα, ε, ποδηλατόδρομοι, ε, όλα αυτά που αναφέρετε είναι πολύ ωραία αλλά λίγο τοπικά. Πρέπει να αξιολογήσουμε Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν κοντά στο σπίτι, στο σπίτι τους. Ε, είναι πολύ δύσκολο νομίζω να μεταφέρουμε τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι. Αυτά είναι λίγο τοπικά λοιπόν που λέτε εκεί. Ε, κατά τα άλλα συμφωνώ ότι η... τα φορτία θα πρέπει να πάψουν να μεταφέρονται οδικώς και θα πρέπει όλο και περισσότερο να μεταφέρονται σιδηροδρομικώς. Συμφωνώ με αυτό. Θα ήθελα να παρουσιάσω μία τροπολογία όπου θα καλέσω την Κομισιόν να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να άρουν τους τοπικούς φραγμούς που αναγκάζουν τα, φορ... τα φορτία να μεταφέρονται οδικώς. Ε, στην, ε, υπάρχει ένας, ένας άξονας Γένοβα-Ρότερνταμ ενδιαφέρει και το Πιεμόντε και τη Λιγκούρια, ε, αυτό, αυτή η πρωτοβουλία μπλοκάρεται ε, και από ε, ένα σημαντικό, μια σημαντική ομάδα των πρασίνων και των αριστερών που εκπροσωπούνται και στο Πιεμόντε, υπάρχουν και στο Πιεμόντε και στη Λιγκούρια. Ε, εγώ ήμουνα δημοτικό σύμβουλο 9 χρόνια ε, πριν έρθω εδώ. Επομένω, τα τελευταία χρόνια ε, ξέρω πολύ καλά τι μάχε δόθηκαν ε, από αυτή την πολιτική, τι πολιτικέ ομάδε. Ε, δεν θέλουν λοιπόν να υλοποιηθεί το τέρτσο βάλικο. Θα πρέπει να υλοποιηθούν αυτά, αυτοί οι άξονε. Θα πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα για την υλοποίηση αυτών των αξώνων. Γιατί αλλιώς η Ιταλία κινδυνεύει να είναι πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ε, μιλάω για τον διάδρομο 5 και το διάδρομο 24. Ε, και κάτι άλλο που ο συνάδελφος μου όχι ο προηγούμενος, ο προπροηγούμενος, που ήθελε να συμπεριλάβει και τις θαλάσσιες μεταφορές και τις εναέριες μεταφορές. Ε, σε αυτό το ψήφισμα που εμείς καταψηφίσαμε, ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Θα ήταν αρνητικό αν ε, συμπεριλαμβάναμε και αυτές τις μεταφορές. Νομίζω ότι ε, σας, έχει, σας έχουν ενημερώσει οι ενέργειες ε, μεταφορές, οι εταιρείε ενέργειων μεταφορών, οι οποίες θεωρούν ότι θα διπλασιαστεί το κόστος τους διπλασιασμός του κόστους τι σημαίνει, διπλασιασμός των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων και προφανώς και των θαλάσσιων εισιτηρίων. Επομένως προσοχή, γιατί εμείς εκπροσωπούμε και τους πολίτες. Γιατί κάποιες επιλογές μας που είναι θετικές για τον περιβάλλον και για την υγεία, τελικά μπορούν να επιβαρύνουν απίστευτα τα πορτοφόλια των καταναλωτών, οι οποίοι κάπως πρέπει να μετακινηθούν παρόλα αυτά. Σας ευχαριστούμε. Αλλά Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με την επιθυμία σας να έχουμε ένα κόσμο που δεν θα έχει τέτοιο βάρος ρήπανσης, δεν θα είναι μολυσμένος. Δεν θέλω να περάσω παράγραφο να παράγραφο, βέβαια, αλλά είναι ένα πρόβλημα το ότι εμείς ασχολούμαστε και πάμε με ποδήλατο ή με τα πόδια στα, στη δουλειά μας. Άλλοι όμως ε, δεν είναι δυνατόν να έχουν ε, τα εμπορεύματά τους σιδηροδρομικά. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου προσπαθούμε το μετρό και τα λεωφορεία και μέσα μαζικής μεταφοράς να έχουμε. Όμως αληθεύει. Πραγματικά είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε πρακτικές, εφικτές λύσεις, ιδιαίτερα για τις διασυνοριακές μεταφορές πρέπει υπό το 7 να κάνουμε κάτι και να πούμε κάτι. Και έχετε δίκιο ότι πρέπει να υπάρξει έρευνα και ανάπτυξη, ώστε οι μικρές κοντινές μεταφορές να αναπτυχθούν και να έχουμε και το θέμα και των εκπομπών ε, που θα μειωθούν. Όπως ο Ματίας και άλλοι είπαν, είναι σωστό η δεύτερη γενεά των βιοκαυσίμων να προαχθεί και να αναπτυχθεί ώστε επιτέλους ε, τα φορτηγά στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους να μην ρηπαίνουν πια τόσο πολύ όπως σήμερα. Το κάνουν αυτό και στο μέλλον θα έχουμε σε λίγα χρόνια διπλασιασμό των όγκων μεταφορών στους δρόμους μας. Ευχαριστώ. Ο Γιώνας έχει τον λόγο παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα να σα πω Συμφωνούμε με τις οκτώ επιμέρους προτάσεις του κυρίου ε, Πρόεδρου. Με αυτές τις συστάσεις, όπως θέλετε να τις ονομάσετε. Υπάρχουν όμως ε, δύο σημεία όπου ο κύριε Λάινεν δεν σταθήκατε αρκετά. Όμω θα πρέπει να τα εξετάσουμε καλύτερα γιατί αποτελούν τμήμα τη πρόταση τη Κομισιόν. Δηλαδή στο 2 παράγραφο 9 εκεί που αναφέρει τα ε, διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Λέει ότι το 1 τρίτον των επενδύσεων ήδη έχουν γίνει. Όμω, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ακόμα απομένουν ακόμη περισσότερο για να γίνουν στο μέλλον. Οπότε θα πρέπει να κάτσουμε και να τονίσουμε τι είδου προσπάθειε πρέπει να καταβληθούν. Πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσουμε στην, προς την υλοποίηση του βορειοανατολικού διαδρόμου. Γιατί υπάρχουν διαφορετικέ πρωτοκαθένες και δικέ του προτεραιότητε. Όμω, θα πρέπει πιο προσεκτικά να λάβουμε υπόψη το ότι έχουν γίνει κινήσει προπαρασκευή επί πολλά χρόνια και υπάρχουν ένα σωρό επιχειρήματα για τον διάδρομο Βόρα Νότου και υπάρχουν επίση πάρα πολλέ χώρε ε, που εμπλέκονται ε, Γερμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ιταλία. Ο δε διάδρομος αυτός είναι θέμα καυτό, επίγει. Είναι κάτι που θα γίνει, θα πρέπει να γίνει για το συμφέρον όχι μόνο των χωρών που προανέφερα, αλλά όλη τη Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να αναχθεί σε ζήτημα υψή τη προτεραιότητα. έχουμε τη γνώμη των ειδικών που καταλήγουν στο ίδιο. Κάτι άλλο τώρα, που δεν είναι άσχετο με το προηγούμενο, η Δυτική Ευρώπη διαθέτει αρκετά προχωρημένο δίκτυο συγκοινωνιών. Είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό το δίκτυο αυτό να επεκταθεί προς Νότο και προς Ανατολάς. Το δε τρίτο κεφάλαιο αυτής της ανακοίνωσης φύγει τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε σαν ένωση στο μέλλον. Αναφέρεται η Βόρεια Αφρική, αναφέρεται ο αυξημένος όγκος των μεταφορών που θα προκύψει και είναι εξίσου σημαντικό να δούμε τι θα γίνει στα Βαλκάνια. Ήδη, εκεί η διαμετακόμιση είναι ένα θέμα καυτό, σημαντικό και θα γίνει ακόμη πιο σημαντικό στο μέλλον. Άρα θα, πρέπει να έχουμε κινήσεις σε επίπεδο ένωσης, θα πρέπει να έχουμε και αντίστοιχη χρηματοδότηση για να προχωρήσουμε. Γιατί, επαναλαμβάνω, το πρόβλημα πρόκειται να γιγαντωθεί την επόμενη δεκαετία κύριε Λάινεν. Αναφέρεται συγκεκριμένα τις αστικές μεταφορές ε, στο σημείο 2, στην πρόταση 2. Το πρόβλημα εδώ δεν μπορεί να λυθεί μια μέρα στην άλλη, αλλά κάτι μπορεί να γίνει να βελτιωθούν τα πράγματα. Και είπαμε ότι πάνω από 80% των Ευρωπαίων ζουν σε μεγάλες πόλεις. Αυτή η τάση φυσικά και μπορεί να αναστραφεί, αλλά μπορεί να συγκρατηθεί. Να ενθαρρύνουμε τον κόσμο που είναι στην Ήπεθρο να μείνει στην Ήπεθρο. Να μην την εγκαταλείψει για να τρέξει στις πόλεις. Βέβαια εδώ και θέμα απασχόληση άμα δεν έχουν δουλειά στην Ήπεθρο τότε τι να κάνουν. Θα πρέπει να έχουν κάποιες ευκαιρίες για απασχόληση. Άρα θα πρέπει και αυτόν τον δείξουμε σε υψηλή προτεραιότητα. Και στην Ανατολική Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία. Θα λύσει έτσι πολλά ε, προβλήματα που έχουν οι πόλεις. Άλλο τώρα που επίσης ε, σχετίζεται με το προηγούμενο, οι μεγάλες πόλεις έχουν πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης των δράσεων που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Οπότε, εάν έχουμε κάποια δίκτυα μεταφορών τα οποία συνδέουν τις πόλεις μεταξύ τους, τις αστικές περιοχές ευρύτερα. Εάν έχουμε επομένω ε, συγκρίσιμες τιμές, συγκρίσιμα κόστη, τότε θετικό είναι το στο πρόβλημα των πόλεων. Και μέχρι σήμερα η Ένωση χρηματοδοτεί έργα υποδομής κυρίως. Δηλαδή, είναι σωστές οι σημερινές ε, προτεραιότητες, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα φρεσκάρουμε, πώς θα αναβαθμίσουμε την υπάρχουσα υποδομή. Και αυτό να το προσέξουμε κυρίως για την κεντρική Ευρώπη. Μια που την δεκαετία του 60 είχαμε υποδομή που αντιστοιχούσε στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Όμως, την δεκαετία του 70 τα πράγματα ε, δεν συνεχίστηκαν τον ίδιο ρυθμό, έγινε απαρχαιωμένη αυτή η υποδομή που τώρα χρειάζεται στις χώρες αυτές. Χρειάζεται. Χρειάζεται καινούργια υποδομή, αλλά τα έργα υποδομής επίσης τα παλιότερα θα πρέπει να τα φροντίσουμε, γιατί αυτό θα προσωπεύει σημαντικές οικονομίες. Διάφοροι συνάδελφοι τόνισαν το πόσο σημαντική είναι η έρευνα και η ανάπτυξη. Αυτά τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο υπαριθμών 7 των το, το, το, όσων μας ανέπτυξε ο Πρόεδρος. Εγώ θέλω πρόεδρε να τονίσω το εξή. Πάνω σε αυτό που αναφέρει. Ότι θα απαιτηθεί συγχρηματοδότηση από την Ένωση και από το κάθε κράτος μέλος για να έχουμε έρευνα για ανάπτυξη ή στα δίκτυα. Συγχρηματοδότηση. Και εν τέλει για το 8 Η πρωτοβουλία που εκεί αναφέρεται είναι κάτι που δεν γνώριζα. Δεν ξέρω τι, με τι πνεύμα διαπνέεται, πάντως μου φαίνεται θεμητή και όπως ε, λέτε σωστά πρώτα θα πρέπει να έχουμε ανταλλαγή των αρίστων πρακτικών, τα κρατη πολύ σωστή αυτή η πρόταση. Και να σας πω από την ε, Ουγγαρία ένα παράδειγμα. Είναι τραγική κατάσταση όσον αφορά τι ε, δημόσιε κοινωνίε στην, στην, στην Ουγγαρία. Υπάρχουν τεράστιε ζημίε που έχουν εσωρευτεί. Όμω, στη δεύτερη πόλη, στον Ντέμπριτζεν, εκεί ε, έχουν φτιάξει ένα δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών που είναι πιο σύγχρονο. Ένα δίκτυο συγκοινωνιών που αντιστοιχεί στις προσδοκίε του κόσμου και χρηματοδοτείται από τις τοπικές αρχές. Να ένα παράδειγμα ε, καλής άριστης πρακτικής που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη και μαζί με άλλες θα μπορούσαμε να τις βάλουμε σε ένα website και να χρησιμεύσει αυτό στις πόλεις που έχουν προβλήματα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε κύριε Άντερ όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στα κρατήδια και στις χώρες έχουμε καλά παραδείγματα για τις μεταφορές. Έχουμε και αρνητικά παραδείγματα. Κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε αυτή η ανταλλαγή να ενδυναμωθεί, ώστε να μάθουμε από τις καλύτερες πρακτικές και να μιμούμαστε τα καλύτερα μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων. Η Σαμπίνα Β. παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας κύριε Λάινεν. Μπορώ να συμφωνήσω σε πολλά τμήματα και υποστηρίζω και τις προτάσεις. 28% έχουμε αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα από το 1990 έως το 2006. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό αναγκαία είναι η μετάθεση των μεταφορών από τις οδικές μεταφορές στις σιδηροδρομικές μεταφορές, ιδιαίτερα των εμπορευμάτων, των αγαθών. Χρειαζόμαστε μια συνολική προσέγγιση για τα σιδηροδρομικά δίκτυα στην Ευρώπη και για το πρόγραμμα διαχείρισης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή κονδύλια στην Γερμανία πάνε για την ανάπτυξη του ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μπαταρίες. Μπορώ να φανταστώ ότι το ίδιο γίνεται και σε άλλες χώρες. Με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχουμε μια μελέτη που πραγματογνωμοσύνη που δώσαμε εντολή να συνταχθεί από πλευρά τη ε, ΓΚΟΕ και δεν θα έχουμε τα επόμενα πέντε χρόνια κάποια μείωση εκπομπών που να αναμένεται από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μπαταρίες. Το αντίθετο θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, αύξηση. Αυτή τη στιγμή η ηλεκτροκινητικότητα χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της εικόνας των ηλεκτροπαραγωγών εταιριών Χρειαζόμαστε όμως ε, κίνητρα για την κινητικότητα μέσω σιδηροδρόμων. Ίσως αυτό στην έκθεσή σας θα έπρεπε να αναφέρετε με σαφέστερο τρόπο και θα υποβάλω και μια αντίστοιχη τροπολογία εγώ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ο Θεόδωρος Κυλακάκης παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, αναφερθώ όχι στα σημεία που συμφωνώ που είναι στο μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της του σχολιασμού, αλλά στο κομμάτι στο οποίο διαφωνώ που αφορά ε, την σχέση μεταξύ ε, ναυτιλίας και χερσαίων μεταφορών. Εδώ πέρα υπάρχει πρόταση να, περιληφθεί, να περιληφθούν οι, ε, οι μεταφορές μέσω ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό Emission Trading System στο σύστημα εμπορίας. Και να γίνει αυτό μόνο για αυτού του είδους τις μεταφορές. Ενώ ξέρουμε ότι οι χερσαίες μεταφορές έχουν πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση από πλευράς ε, CO2. Ξέρουμε επίσης ότι οι χερσαίες μεταφορές άλλες εντάσσονται στην πραγματικότητα στο σύστημα και άλλες δεν εντάσσονται. Δηλαδή έχουμε το τρένο το οποίο κινείται με ηλεκτρισμό κατά συνέπεια εντάσσεται στο σύστημα μέσω της ηλεκτρικής ενέργειας την οποία καταναλώνει και έχουμε όλες τις οδικές μεταφορές οι οποίες είτε είναι εμπορευματικές είτε είναι για μετακίνηση ατόμων ε, επιβατών δεν εντάσσονται στην πραγματικότητα στο σύστημα και οι οποίες γράφουμε στο ίδιο μέρος ότι αυξάνονται δραματικά. Τι θα συμβεί λοιπόν αν βάλουμε μόνο τις μεταφορές ναυτιλίας στο σύστημα. Καταρχήν θα ενθαρρύνουμε τη μετα... την... Μετα... τις μεταφορές της χερσαίας εις βάρος της ναυτιλίας, ενώ ξέρουμε ότι η ναυτιλία είναι πιο φιλικά περιβαλλοντική σε ό,τι αφορά το CO2 τουλάχιστον και από αρκετές άλλες πλευρές. Δεύτερον, θα ενθαρρύνουμε, εφόσον μιλάμε μόνο για ευρωπαϊκό σύστημα, σε εμά στην Ελλάδα για παράδειγμα, να αντί να έρχονται τα πλοία στα δικά μας λιμάνια, να πηγαίνουν στα διπλανά λιμάνια της Τουρκίας και να μας έρχονται με φορτηγά, τα οποία θα περνάνε από την Ελλάδα, τα εμπορεύματα για να πάνε είτε στη χώρα μας, είτε στην υπόλοιπη Βαλκανική, είτε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε δηλαδή πολύ συγκεκριμένο carbon leakage, άλλες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, οι οποίες δεν μπορεί να, τις, να διαφορούμε για αυτές. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια πιο σύνθετη προσέγγιση, η οποία αναλαμβάνει υπόψη το σύνολο του τομέα των μεταφορών. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ένα καράβι που μεταφέρει χιλιάδες τόνους από ένα εμπόρευμα είναι κοινωνικά λιγότερο χρήσιμο από μία BMW που τρέχει με 200 χιλιόμετρα σε μία οτοστράτα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα έχουμε στο ψήφισμα για τις κλιματικές αλλαγές για την Κοπενχάγη είπαμε ότι στις ναυτιλιακές μεταφορές και στις εναέριες μεταφορές μια σφαιρική συμφωνία στοχεύουμε να πετύχουμε να υπογραφεί ώστε να αποφύγουμε στρεβλώσεις ανταγωνισμού. Εντάξει, παρακαλώ τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Σταμάτο, να τοποθετηθεί σε αυτό το θέμα, μας πει δύο λόγια. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα διάφορα θέματα να αναφέρονται, τα οποία σχολιάζει και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι υπάρχει μια ευρεία λοιπόν συμφωνία για πολλά από αυτά που αναφέρατε άκουσε να λέτε, Φερρυπίν, πολύ το είπατε μάλιστα, ότι η εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους είναι σημαντικό πράγμα. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και κατέχει κύρια θέση στην ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια βιώσιμη για βιώσιμες μεταφορές με μικρότερο, με μικρότερες εκπομπές. Η έρευνα και η ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αν δείτε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήδη στον τίτλο, από τον τίτλο μπορείτε να καταλάβετε τι θεωρούμε ότι είναι οι βασικές, ποιες είναι οι βασικές ε, προτεραιότητες, οι τρεις βασικές προτεραιότητες. Καταρχάς είναι η ενσωμάτωση των διαφορών τρόπων μεταφορών, Κάτι που σκοπεύει να δώσει και κίνητρα να φύγουν πολλές μεταφορές από το δρόμο για να προωθήσουμε άλλες μεθόδους μεταφορών πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο που θα διευκολύνει και την κινητικότητα και δίνει και καλές υπηρεσίες στους χρήστες. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η τεχνολογία. Και εδώ υπάρχουν διαφορετικές ε, τεχνολογίες σε διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης. Κάποιος μίλησε για τα βιοκαύσιμα. Ε, θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή λύση ε, για κάποιες, ε, κάποιους τρόπους μεταφορών. Παραδείγματο χάρη για την αεροπορία, όπου άλλες λύσεις είναι πιο δύσκολες να εφαρμοστούν. Φυσικά υπάρχει, υπάρχουν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, Υπάρχουν και άλλε τεχνολογίες που είναι λιγότερο ανεπτυγμένε ακόμα και πολύ πιο μακριά από την αγορά, αλλά μπορούσαν να, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Η άποψη τη Κομισιόν είναι ότι θα πρέπει να κρατήσουμε μια κάποια τεχνολογική ουδετερότητα και ταυτόχρονα να προσφέρουμε σε άλλες ε, τεχνολογίες, ε, είτε τις υποδομές ε, ή προγράμματα επίδειξης για τεχνολογίες που είναι λιγότερο ανεπτυγμένε. Κάποιο άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό για την ανακοίνωση, ε, το τονίσατε λιγότερο εσείς οι βουλευτές, είναι το θέμα των χρηστών. Θα δείτε ότι στην ανακοίνωση υπάρχει όρος φιλικός προς τον χρήστη. Αυτή είναι μια ευρεία έννοια, που καταρχάς σημαίνει ότι θα πρέπει να προσφέρουμε ασφαλείς μεταφορές στους χρήστες. Αλλά για να έχουμε και αλλαγές στις συμπεριφορές των χρηστών και στον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα μεταφορών, θα πρέπει να δώσουμε ποιοτικέ υπηρεσίες και βιώσιμες εναλλακτικέ λύσεις στους χρήστες. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπάρξει μια αλλαγή. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες. για τον θαλάσσιο και αέριο τομέα που τον αναφέρατε. Ένα σχόλιο. Η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτοί οι δύο τομείς μεταφορών θα πρέπει και αυτοί να συνεισφέρουν για τη, στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Είναι δύο τομείς διεθνείς, επομένως είναι εκτεθειμένες, στο διεθνή ανταγωνισμό Υπάρχει το πρόβλημα να δοθούν σημαίε ε, σε άλλα πλοία στο εξωτερικό, στον, στην αυτιλ, στον αυτιλιακό τομέα. Υπάρχει και, το, και ο κίνδυνο της διαρροής του διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να βρεθεί μια παγκόσμια λύση για αυτού του δύο τομείς. Γι' αυτό ακριβώς η διαπραγματεύση σε διεθνή βήματα ε, είναι να εξελίξει. Και όταν μιλάμε για παγκόσμια λύση, Φυσικά έχουμε υπόψη μας ε, ένα εργαλείο με βάση την αγορά, που θα μπορούσε να είναι το ETS ή θα μπορούσε να είναι ένα τέλος στα καύσιμα. Νομίζω ότι αυτά αρκούν από μέρους μου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αμάτο. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα αυξηθούν οι όγκοι μεταφορών τα επόμενα δέκα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα δώσει πρόσθετα προβλήματα και είναι έργο των πολιτικών και της πολιτικής αυτή την αρνητική εξέλιξη να την επανορθώσει και να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις. Και γι' αυτό η Νέα Λευκή Βίβλος και ο προπομπός αυτής, αυτή, αυτή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από τη Λευκή Βίβλο. Υπάρχει συνένεση που διαπιστώνω στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή η κατάσταση όσον αφορά τον ανταγωνισμό διεθνώ αναφέρθηκε από εσά όσον αφορά τι ναυτιλιακέ μεταφορές γιατί είμαστε πιο θαραλέοι στι ενέργειε μεταφορέ. Έχουμε ήδη συμπεριλάβει στο σύστημα εμπορία τρύπων τις ενέργειε μεταφορές. Πρέπει να δούμε τώρα τι θα γίνει με τις ναυτιλιακέ μεταφορές. Πώς θα μπορέσουν αυτέ να ενταχθούν και με ποιο τρόπο. Η επιθυμία για κινητικότητα είναι κάτι που είναι ανθρώπινη ανάγκη δεν νομίζω ότι μπορεί να απαγορευτεί η κινητικότητα των πολιτών. Όμως παρόλα αυτά μπορεί να οδηγηθεί σε σωστού διάβλους και να χειραγωγήσουμε με σωστό τρόπο αυτή την κινητικότητα. Υπάρχουν καλά παραδείγματα ενός model split, ενός προτύπου που θα ακολουθείτε και θα υιοθετείτε που θα είναι καλύτερο όσον αφορά τις μεταφορές και την κυκλοφορία στα αστικά κέντρα και να μην υπάρχει αποτελμάτωση και συμφόρηση εκεί. Υπάρχει μια διαφορά βόρειων και νότιων χωρών σε αυτό το θέμα και στις ίδιες τις χώρες κιόλας στην επικράτειά Στο βορρά φαίνεται αυτό το modal split, η διαφορετική χρήση διαφορετικών φορέων να χρησιμοποιείται με καλύτερο τρόπο με περιορισμούς ε, για την πρόσβαση στα αστικά κέντρα, στον πυρήνα των πόλεων, με μια προσφορά ποδηλάτων για ποδηλατοδρόμους ε, και χρήση ποδηλάτων. Είχα πάει με την αντιπροσωπεία στη Στοχόλμη και εξεπλάγει ότι υπήρχε δημόσια, υπήρχαν δημόσια, ε, δημόσια σταθμοί ε, για να φουσκώσει κανείς ε, με αέρα τα λάστιχα του ποδηλάτου του. Η δημόσια υπήρχε προσφορά ποδηλάτου για κάποιον που είχε πρόβλημα με το λάστιχό του. Είναι ένα στοιχείο λοιπόν αυτό ένα στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει. Δεν κοστίζει πολλά. Αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα μπορεί να βοηθηθεί άμεσα με ένα τέτοιο τρόπο. Αυτή η ανταλλαγή λοιπόν αναμεταξύ μας των βέλτιστων πρακτικών θα έπρεπε να διοργανωθεί σε ευρύτερο πλαίσιο και να προαχθεί και με την Επιτροπή των Περιφερειών όπου οι περιφέρειες και οι δήμοι και οι κοινότητες εκπροσωπούνται μπορούμε να διοργανώσουμε θετικές τέτοιες ε, εκδηλώσεις και μέτρα. Όχι μόνο στην ίδια την πόλη, αλλά και πέρα στην Ήπεθρο και είναι θετικό να υπάρχει χρήση αυτού του προτύπου ε, όσον αφορά την θετική χρήση των μέσων μεταφορών ε, στην πόλη και να επεκτείνονται στο, στην Ήπεθρο. Δεν είναι καλό να μην υπάρχει προς την Ήπεθρο δίκτυο και να είναι αναγκασμένοι όλοι να χρησιμοποιούν το ταχύ τους. Πρέπει να υπάρξουν καλές προσφορές λοιπόν μέσα σε αυτή τη διαδικτύωση Τώρα, βιοκαύσιμα, ευρωβινιέτα, καλές ιδέες ε, που πρέπει να ενταχθούν εδώ στην έκθεσή μου, στο σωστό σημείο. Αν θέλουμε και τις ιδεοδρομικές μεταφορές να τις προαγάγουμε, έχουμε μεγάλες ελλείψεις σχετικά με αυτό στην Ευρώπη. Η τεχνολογία δεν είναι η καλύτερη στους ιδεοδρόμους μας και κυρίως η πανευρωπαϊκή σιδηροδρομική πολιτική χωλαίνει πίσω από τις προσδοκίες των πολιτών. Αναφέρθηκαν οι διάδρομοι corridors βορρά-νότου και από τον βορρά προς Ανατολάς. Υπάρχουν τόσες πολλές αντιστάσεις όμως και δημιουργούνται τριβές, εν μέρη κιόλας και κρατικών επιχειρήσεων σιδηροδρόμων ε, οργανισμός Σιδηροδρομικών Μεταφορών. Αντιστάσεις λοιπόν που παρακολύουν, παρεμποδίζουν να έχουμε μια πραγματική απρόσκοπτη ε, διεξαγωγή μεταφορών. Θα έλεγα οι μεταφορές αγαθών από την Σκανδιναβία για, προς την Ισπανία αντιμετωπίζουν ε, ασύλληπτα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει κανείς και ελπίζουμε ότι στη νέα περίοδο προγραμματισμού θα γίνει μια νέα κίνηση θα κερδίσουμε με μια νέα αφετηρία. Γιατί διαφορετικά είναι κρίμα να έχουμε τέτοιε επιθυμίε και προσδοκίε και να μην γίνεται τίποτα. Πρέπει η Ευρωβουλή να προσέχει περισσότερο οι αποφάσει ε, να τηρούνται και να εφαρμόζονται, να εκτελούνται. Υπάρχει έλλειμμα που πρέπει να καλυφθεί. Θα έλεγα λοιπόν ότι συμφωνώ με πολλά που ε, προαναφέρατε εσείς συνάδελφοι στα σχόλιά σας. Ελπίζω στη συνέχεια ότι θα καταθέσετε τροπολογίες για αυτά τα αιτήματά σας. Θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, προθεσμία για την κατάθεσή τους. 12 το μεσημέρι, 9 Δεκεμβρίου προσδοκώ αυτά τα οποία είπατε να κατατεθούν με μορφή τροπολογιών, ώστε να έχουμε μια θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή μας που θα διαβιβάσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών. Ευρωπαϊκές μεταφορές μέχρι το 2020 είναι μεγάλο χαρτοφυλάκιο, πολύ ε, περίπλοκο θέμα και όσον αφορά την ημερήσια διάταξη γι' αυτό. Τώρα λοιπόν ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση σε αυτό το σημείο. Ή η κυρια Ντεμπρόιν έχει μία παρατήρηση. Εσείς κυρία Ντεμπρόιν, παρακαλώ. Uh, δεν ξέρω αν άκουσα καλά τη διερμηνία. Μιλήσατε για τις 19 Δεκεμβρίου. Λυπάμαι. 9 Δεκεμβρίου, 9 Δεκεμβρίου είναι, 12 το μεσημέρι προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Σας ευχαριστώ. Το τελευταίο σημείο ήταν εκείνο που είχε απομείνει από εχθές, το υπαριθμό 5, μια στιγμή. Ναι. Η έκθεση Ρόσμπαχ λοιπόν. η κυρία Ρόσμπαχ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη για το θέμα μου. Τον Οκτώβριο ήδη 1990 άκουσον άκουσον υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια κράτη-μέλη και κάποια γειτονικά κράτη μια συμφωνία υπέγραψαν ώστε από κοινού να αντιμετωπιστεί η ρήπανση του βορειοανατολικού Ατλαντικού. Πρόκειται εδώ για μια ολόκληρη σειρά συμβάσεων. Πρόκειται για τη σύμβαση του Ελσίνκη, για την σύμβαση της Βόνης για τη Βόρεια θάλασσα, θάλασσα και ε, βλαπτικές ουσίες. Επίσης για την σύμβαση της Βαρκελόνης και φυσικά πρόκειται πάλι επίσης για τη Μεσόγειο. Υπάρχει και μια σύμβαση της Λισαβόνας πόσο αφορά την Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο, Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τον Οκτώβριο 1990 υπεγράφει. Αλλά λόγω ενός επίμαχου θέματος επικράτη, δικαιοδοσίας ε, μεταξύ Μαρόκο και, Μαρόκου και Ισπανίας για τη Δυτική Σαχάρα. Δηλαδή δεν υπεγράφει, δεν επικυρώθηκε. Τώρα, μετά από πολλά χρόνια, μετά από 20 χρόνια, η Ισπανία και το Μαρόκο κατάφεραν να συμφωνήσουν. Και υπήρξε ένα πρόσθετο πρωτόκολλο το οποίο από την Πορτογαλία και την Γαλλία προσυπεγράφει. Και σε αυτό αναφερόμαστε τώρα και γνωμοδοτούμε γι' αυτό. Η Συμφωνία λοιπόν Σύμβασης Λισαβόνας αφορά την πρακτική συνεργασία, πρακτική μορφή συνεργασίας. Τι θα κάνουμε όταν υπάρχει μεγάλη ρήπανση μεγάλης κλίμακας των θαλασσών μας ή των περιφερειών μας. Προσπάθησα να διαβάσω το δυνατόν περισσότερα κείμενα σχετικά ώστε να εξοικειωθώ. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ λογικές οι διατάξεις αυτής της σύμβασης και ότι επιτέλους ήρθε η χρονική στιγμή να προωθήσουμε μια τέτοια συνεργασία και να την εφαρμόσουμε χειροπιαστά. Κάνουμε λόγο εδώ για μια περιφέρεια που επεκτείνεται από τις Αζόρες μέχρι την ε, βορειοανατολική Ευρώπη. Είναι θαλάσσιες οδοί με μεγάλη πυκνή κίνηση όσον αφορά τις μεταφορές. Ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν έχει εξεταστεί προσεκτικά, το οποίο όμως θα ήθελα να αναφέρω εδώ, είναι τα πλαστικά τα οποία κυκλοφορούν στους, ε, στις ε, θάλασσές μας είναι κάτι που είναι σε, έχει έκταση 34 φορές μεγαλύτερη από την επικράτεια της ε, Ολλανδίας. 34 φορές μεγαλύτερη από το εμβαδόν της ε, Ολλανδίας αυτή η ε, πλαστική θάλασσα, ας το πω έτσι, με πλαστικά προϊόντα. Κάτι πρέπει να κάνουμε το δυνατόν γοργότερα, Πρόεδρε. Μάλιστα, σωστό, πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ιδιαίτερα για εκείνους που ζουν στις παράκτιες περιοχές, αλλά και για τα έμβια όντα που ζουν στη θάλασσα, στις θάλασσες αυτές, σίγουρα. Η κυρία Ντεμπρόιν ήταν στον κατάλογο, έχετε τον λόγο. Μία ερώτηση, κυρία Ρόσπαχ. Αναφέρατε συγκεκριμένα, κυρία Ρόσπαχ, ότι η Πορτογαλία, η Γαλλία και οι υπές χώρες έχουν τώρα υπογράψει. Και μιλάω για το θέμα της Δυτικής Σαχάρας φυσικά. Θα ήθελα να μας ξεκαθαρίσετε, εάν οι εκπρόσωποι του λαού της Δυτικής Σαχάρας έχουν δεχθεί τη θέση αυτή, την οποία μας παρουσιάσατε. Καθότι, από γνωρίζω από, από ξέρω... ναι. Καθότι γνωρίζω τα ναι. έγινε δεκτό από το Μαρόκο. Το 2008 υπεγράφει. Και από το Μαρόκο, λοιπόν, λέει η κυρία Ροσμπαχ. Δηλαδή πρέπει να απαντήσω στο ερώτημά σα με ναι. Το Μαρόκο είπε ναι. Δεν είναι το ίδιο όμω η Σαχαράουι με το Μαρόκο. Αυτή ήταν η ερώτηση. Οι κάτοικοι τη Δυτική Σαχάρα, μάλλον δεν έχουν λέγει, δεν έχουν δική του ε, θέση, δεν επετράπει να διατυπώσουν τη δική του φωνή να διατυπώσουν τη δική του φωνή για την Δυτική Σαχάρα. Οι Σαχαράουι, αν θα έχουν φωνή στη διεθνή κοινότητα για τέτοια θέματα, αμφιβάλλω γι' αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, δεν έχουμε άλλους που να ζητούν τον λόγο. Και εδώ έχουμε προθεσμία για τις τροπολογίες 9 Δεκεμβρίου, 9 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Εντάξει. Και περνάμε στο σημείο 18. Διάφορα. Υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει τίποτα. Ήταν η τελευταία μας συνεδρίαση εφέτος λοιπόν αυτή. Στις 25 Ιανουαρίου θα ξανασυναντηθούμε πιθανότατα για τις ακροάσεις των επιτρόπων, νέων επιτρόπων. Θα πρέπει αυτό να διακριβωθεί στη συνέχεια. Αν θα συμμετάσχουμε και πώς. Όταν θα υπάρχουν πλέον νέα στοιχεία. Λίγη συνεδρίασή μας. Σας εύχομαι καλό τέλος 2009 και καλές γιορτές.